με το θέμα Οικονομική Διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα δώσω μέσα το λόγο ξανά στον κύριο Αντιπρόεδρο Κατάινεν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Είναι ένα από τα θέματα στα οποία συνεργάζομαι και με άλλους συναδέλφους στην Επιτροπή όπως επίσης και με την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη και προσπαθούμε ακριβώς να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική την οικονομική διπλωματία. Χρησιμοποιούμε δηλαδή όλους τους μοχλούς που έχουμε στη διάθεσή μας ε, στα πλαίσια της οικονομικής μας δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει απομάκρυνση εμποδίων, κίνητρα για το εμπόριο άνοιγμα διεθνών αγορών. Διακανονιστική και ρυθμιστική σύγκληση, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία υποστηρίζουν την διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης μας. Η οικονομική διπλωματία είναι λοιπόν στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας που κάνουμε για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Βασική δηλαδή προτεραιότητα του προγράμματος Juncker. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα και τους μοχλούς που έχουμε στη διάθεσή μας για να προωθήσουμε την ευμάρεια της Οικονομικής Ένωσης και των πολιτών της. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια πιο συνεκτική ε, πολιτική που να ελέγχει τις οικονομικές εξελίξεις χρησιμοποιώντας ε, τις επενδυτικές μας δυνατότητες και τις αναπτυξιακές μας προσπάθειες. Η εξωτερική πολιτική έχει μία σαφέστατη βέβαια οικονομική διάσταση και θα πρέπει η πρόσβαση στη χρηματοδότηση ε, κάποιων επιχειρήσεων για εξαγωγές να ενισχυθεί οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εργάζονται προς την κατεύθυνση της απόσυψης των εμποδίων και ανοίγοντας τις, φερικές, τις ε, παγκόσμιες αγορές, προωθώντας την διακανονιστική σύγκληση και αποκαθιστώντας την δίκαιη εμπορική ε, συναλλαγή. Υποστηρίζουμε επίσης και τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το κάνουμε αυτό διαπραγματευόμενοι ε, ε, εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες χρησιμοποιώντας και διπλωματικά διαβήματα από τις αντιπροσωπείες μας και στα πλαίσια των επαφών υψηλού επίπεδου με άλλες χώρες και αναπτύσσοντας και οικονομικές πρωτοβουλίες για την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων, διευρύνοντας την πρόσβαση στις αγορές, αυξάνοντας τον αριθμό των εμπορικών αποστολών και αυξάνοντας τις εμπορικές συνεργασίες. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερο όμως για να βελτιώσουμε ε, την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στρατηγικών μας στόχων. Και θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική αυτή και σε σχέση με μέσα που θα διασφαλίσουν την συνοχή η ενότητα και ο συντονισμός θα πρέπει να διασφαλιστούν και με το Ευρωκοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη γιατί μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρότερη από ό,τι μεμονωμένα οι χώρες μας. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα και ε, μέσω εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Τράπεζας Επενδύσεων και της Υπηρεσίας Εξωτερικών θεμάτων. Η ομάδα αυτή ήδη έχει βοηθήσει τον συντονισμό μας εσωτερικά. Ένα από τα επόμενα βήματα είναι να εμπλέξουμε τις αντιπροσωπείες που έχουμε τις εμπορικές, να τους δώσουμε καλύτερες οδηγίες. Προσπαθούμε να δούμε επίσης και το πώς θα βελτιώσουμε τον συντονισμό με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Σεβόμενοι επίσης και τις διαδικασίες διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αποφεύγοντας τις επικαλύψεις. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τους τομείς τους οποίους η ευρωπαϊκή δημοκρατία, διπλωματία συγγνώμη, πρέπει να ενισχυθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ρόλος του στα πλαίσια της διπλωματίας είναι κομβικός γιατί έχετε σχέσεις με τα κοινοβούλια των περισσότερων χωρών στον κόσμο. Απαιτείται να πετύχουμε τους κοινού στόχους και να προστατεύσουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα. Θα ναι. σταματήσω εδώ και θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Πρώτος ομιλητής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εξ ονόματος ε, του ΕΛΚ. λεπτό κύριο Σταγιάννη, Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Αν θέλει να παίξει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνέ επίπεδο, πρέπει να προωθήσει την αντιγωνιστικότητά τη μέσω τη βιομηχανία και τη ενέργεια. Και για να πετύχει το στόχο αυτό, θα πρέπει να αποκτήσει πραγματική οικονομική διπλωματία και να έχει συγκεκριμένου στόχου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις τη στο εξωτερικό για να μπορέσει να λάβει θέσεις στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Άπο Ανατολή και να παγιωθεί εκεί. Δεύτερον, να προωθήσει τι πρωτοβουλίε διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω αποστολών σε αναπτυσσόμενες ε, χώρες και B2B. Αυτό είναι το καλύτερο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τη μετακατάσταση των επιχειρήσεών μας. Τρίτον, να προσελκύσουμε επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τουριστικές ροές. Η Κομισιόν ήδη έχει ε, αναπτύξει εργαλεία που υποστηρίζουν αυτές ε, αυτούς τους τομείς. Σκέφτομαι, παραδείγματο χάρη, κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί σε 30 περιφέρειες και έχουν βοηθήσει τι επιχειρήσει σα να επεκταθούν πέρα από τα σύνορα τη Ένωση. Όμω, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να δράξουμε ευκαιρίε σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική ε, δράση. Ε, πρέπει ε, να επικεντρωθούν οι αρμόδιοι στην υποστήριξη των μικρών μα επιχειρήσεων. Όμω δεν έχουμε αναπτύξει τον κατάλληλο προβληματική που θα τι βοηθούσε περισσότερο να αναπτυχθούν. Εμεί θέλουμε να έχουμε έχουμε αποστολές που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ελπίζω όσα είπατε να τα ακολουθήσουν και άλλοι επίτροποι. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Γκραπίνη για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, ε, κυρίες και κύριοι. οικονομική διπλωματία δεν είναι νέα έννοια. Δεν τη συζητούμε εδώ για πρώτη φορά απόψε. Ε, θυμάμαι ε, τις δραστηριότητες του κυρίου Ταγιάννη όταν ε, ήταν αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2013 είχε αρχίσει ο ίδιος ένα πολύ σημαντικό ε, πρόγραμμα για την οικονομική διπλωματία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πρωταγωνιστεί. Η οικονομική διπλωματία είναι εξωτερική πολιτική με πάρα πολύ σαφείς κανόνες και στόχους την προώθηση της οικονομικής ευημερίας των πολιτών μας. Χρησιμοποιεί η οικονομική διπλωματία τα εργαλεία της εξωτερικής πολιτικής για να υποστηρίζει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών των κρατών μελών. Για να επιτύχει αυτό το στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθεί την ανταγωνιστικότητα παγκοσμίω. Θα πρέπει να διατηρεί ή να αναλάβει στρατηγικό ρόλο, σε, ε, ηγετικό ρόλο μάλλον σε στρατηγικούς τομείς. Ο ίδιος ο κύριος Γιούγκερ, ε, λέει ότι θα πρέπει να διεθνοποιήσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο και να υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες. Το είπατε και εσείς αυτό κύριε Επίτροπε, αλλά δεν μας λέτε και πώς θα το κάνετε διότι αν δεν έχουμε και τον προπολογισμό που χρειάζεται για να υποστηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διεθνώς, θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Είναι σαφή η ερώτησή μου και ελπίζω να έχω και σαφή απάντηση. Ποια είναι τα διπλωματικά εργαλεία που σκέφτεστε τώρα να αναπτύξετε τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πάρα πολύ σημαντικές διαπραγματεύσει με μεγάλες αγορές όπως είναι η ΕΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία κλπ. Και ως πρόεδρος του Intergroup για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχω συναντήσει πολλούς, έχω διατελέσει και υπουργό στη χώρα μου μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ποια οικονομική διπλωματία θέλετε να στήσετε λοιπόν για να βοηθήσετε τις μικρομεσαίες να επεκτείνουν τις δραστηριότητε τους σε τρίτες χώρες. Τι μπορεί να γίνει για να είναι πιο καινοτόμες, πιο ισχυρές, πιο παγκόσμιες οι δικές μας μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχετε σχέδιο, έχετε παγκόσμια στρατηγική για παραγωγή ε, πλούτου, για πρόθεση ευρωπαϊκών αξιών με υγεία, ανταγωνισμό. Η οικονομική διπλωματία είναι πάρα πολύ σημαντική διεθνώς και θα αναζωογονήσει την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Από το ECR το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κρασνοντεύσκη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα χρησιμοποιώντα ε, το μέσο της οικονομικής διπλωματίας. Θα μπορούσαμε να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις μας και τα προϊόντα μας. Θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε περισσότερους επενδυτές στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και το θέμα των χωρών και των περιφερειών να γίνονται αυτά σε επίπεδο χωρών και περιφερειών. Το ανέφερε αυτό ο κύριος Κατάινεν, αλλά χρειαζόμαστε και νέους τρόπους και μεθόδους για να διεξαγάγουμε την οικονομική διπλωματία. Αυτή η οικονομική διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των χωρών και των περιφερειών της Ευρώπης. Θα πρέπει να ενδυναμώσει τις ε, δραστηριότητες των κρατών μελών και όχι να τις αντικαταστήσει. Όμως ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Το χάσμα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου και των περιφερειών αυξάνεται. Η οικονομική διπλωματία με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στοχεύει στο να καλύψει αυτά τα κενά και να εξελίψει τις διαφορές. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων, κυρία Σχάκε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Επίτροπε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Γίνεται την κατάλληλη χρονική στιγμή και την υποστηρίζουμε εμείς. Το συζητήσαμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επικεντρωθεί στο εσωτερικό της και τώρα βλέπουμε προς τα έξω και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μόνο απειλές εκεί έξω αλλά και πολλές ευκαιρίες. Ένα από τα ισχυρά σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φυσικά η διπλωματία και νομίζω ότι η οικονομική διπλωματία είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουμε μια σαφή εικόνα για τους ανθρώπους γιατί έχουμε το εμπόριο και τις άλλες οικονομικές πολιτικές και τι μπορούν να σημαίνουν για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα για το ότι πρέπει να έχουμε ένα δρόμο διπλής κατεύθυνσης, ότι έχουμε τους διπλωμάτες μας και τους εκπρόσωπους μας που αναζητούν ευκαιρίες σε τρίτες χώρες, αλλά θα πρέπει να καλωσορίσουμε και όσους ε, φέρνουν και γνώση πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ε, λιγότερο ανταγωνιστικοί παγκοσμίω και να ε, δρούμε από κοινού όλοι μαζί ως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουνα πρόσφατα στην Βοστόνη ως αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας και και είχαμε κάποιες νέες επιχειρήσεις, ε, ένα φυτόριο επιχειρήσεων, είχαμε ένα σουηδικό, γερμανικό κόμβο και λειτουργούσαν πολύ κοντά το ένα στον άλλον. Γιατί να μην ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να δείξουμε τι έχει να προσφέρει η Ευρώπη και να ε, φέρουμε την επιχειρηματικότητα ε, και άλλους παράγοντες ξανά σε επαφή με πρωταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το ίδιο είχε συμβεί και στην περίπτωση τη Silicon Valley. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλέξουμε και την τεχνολογία, να χρησιμοποιήσουμε ε, και την τεχνολογία των πληροφοριών, να εμπλέξουμε τον ιδιωτικό τομέα και αυτοί θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο στο να εφαρμόσουν και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη. Ευχαριστώ. Γκουε, NGL, ο κύριος Σόλτ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτό που μας λέτε ε, για την οικονομική διπλωματία, για την επιρροή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να δημιουργείται ε, νέα αγορά και θα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τομείς, όλα τα θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτά θα πρέπει όμως να απαντηθούν τα ερωτήματα. Τι σημαίνει αυτό. Για να πετύχει το εμπόριο ε, θα πρέπει να είναι μεταξύ ε, ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Αυτό δεν δημιουργεί μόνο ε, νέες αγορές, αλλά προκαλεί και ένα μεγάλο πρόβλημα. 50% του εμπορίου γίνεται μεταξύ χωρών του Νότου πλέον. Ε, που λαμβάνουν υπόψη τα δικά τους συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν το καταλάβει, ε, στο μέλλον ε, θα αποτύχει. Θα πρέπει η εμπορική πολιτική μας να είναι ισορροπημένη, γιατί θα βρούμε το μάστορά μας. Ήδη πάνω από το 1 τρίτο του παγκοσμίου εμπορίου γίνεται στο νότο. Χρειάζεται δηλαδή να το ξανασκεφτούμε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρας έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι αφενός που κατατέθη αυτή η ερώτηση με την ηγεσία του κυρίου Ταγιάννη και τους υπολείπους ε, της ομάδας ε, της διακομματικής για τις μικρομεσές. Ήδη στις 13 Οκτωβρίου του 2015 στο Intergroup Μικρομεσές ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα και χαίρομαι επίσης ε, γιατί η Αυστρία ε, έχει ε, ρόλο ηγετικό, έχει ρόλο πρωτοπόρο με την οργάνωση εξωτερικού εμπορίου μας και έχουμε παρουσία διεθνή με εξαγωγές, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αυστρίας. Το είπατε 80 με 90% της οικονομικής ανάπτυξης ε, τα επόμενα 10 με 15 χρόνια θα γίνεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 1 τρίτο στην Κίνα παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή μόλις 13% όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης δραστηριοποιούνται εκτός της ίδιας της χώρας τους, όχι πόσο μάλλον της Ένωσης και 25% μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδύσεις λοιπόν στην παγκοσμιοποίηση ε, σε μεγάλο βαθμό γίνονται εκτός της Ευρώπης. Θέλουμε να μεταξελίξουμε το ΕΦΣΥ και να συζητήσουμε και για τις χώρες της Αφρικής, για τους γείτονές μου. Ε, οι μικρομεσαίες χρειάζονται καθοδήγηση, βοήθεια, υποστήριξη, να τους ανοίγει κάποιος τις πόρτες γιατί δεν μπορούν μόνες τους. Εξού και η συνεργασία, ε, η οικονομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αυτά όλα θα πρέπει να συνενωθούν. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Φρανσίσκο Ασίς. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, οι οικονομίες είναι όλο ένα και πιο αλληλεξαρτώμενες και επομένως η οικονομική διπλωματία πρέπει να αποτελεί ένα θεμελιώδη φορέα όλων των εξωτερικών πολιτικών. Θα πρέπει να έχει δύο κυρίους στόχους στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αφενός να συνεισφέρει στη διεθνοποίηση ε, του επιχειρηματικού μας ιστού και δεύτερον να προσελκύει ξένες επενδύσεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον πρώτο στόχο να υποστηρίξουμε τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις γιατί αυτές χρειάζονται χρειάζονται περισσότερο την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη είχαν πάρα πολλέ φορές την υποστήριξη των κρατών μελών να χρειάζονται και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχουν δυσκολίες για να κατακτήσουν νέε εξωτερικές οικονομίες. Και ενώ τώρα διαπραγματευόμαστε εμπορικέ συμφωνίε με διάφορε χώρε και ομοδοποίησεις χωρών, αυτή η πρόκληση λαμβάνει μια ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε πολύ συγκεκριμένα μέσα από χρηματοοικονομική σκοπιά μέχρι και την ε, ε, βοήθεια στην επιμιλητή έτσι ώστε να επιτρέψουμε στον επιχειρηματικό μας ιστό ε, για να διεθνοποιηθεί γρηγορότερα και να μπορεί να ανταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο. Η δεύτερη πτυχή είναι πολύ σημαντική και έχει να κάνει με την ικανότητα να προσελκύσουμε καλέ ξένε επενδύσει στον πολιτικό και οικονομικό χώρο τη Ευρώπη. Πολλά μπορούν να γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριο Γιάννο Λεβαντόφσκι για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ αποδέχομαι την διάγνωση όπως επίσης και την συνταγή την οποία προέκρινε ο κύριος Ταγιάννη και ο κύριος Κατάινεν. Προφανώς και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τις δυνάμεις όλων των οργάνων. Θα ήθελα να πάρω το λόγο όμως σήμερα γιατί όπως ακριβώς και ο πρόεδρος, όπως ακριβώς έχω πει σαν πρόεδρος της ε, διακοινοβουλευτικής με το Ιράν. Έχουμε το άνοιγμα μιας τεράστιας αγοράς με πολύ υψηλές δυνατότητες. Τι συνέβη από τότε που υπεγράφει συμφωνία. 144 επίσημες επισκέψεις επισήμων από διάφορες χώρες που ανταγωνίζονται για αυτό το νέο έδαφος. Η προσπάθεια που έχουμε να κάνουμε είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους επενδυτικούς χώρους να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες και να μοιραστούμε σωστή ενημέρωση. Αυτό ε, είναι που κάνουμε σε σχέση με τις 144 επίσημες εμπορικές επισκέψεις και ποιος ξέρει πόσες εκατοντάδες ανεπίσημες. Έχουμε λοιπόν κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Ε, εμείς ε, ε, μένουμε μερικές φορές σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο πολλές φορές κάποιες χώρες δεν δέχονται εύκολα. Ο κύριος Μάρκος Πίπερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πιτροπέ, η ενέργεια και η μεγάλη βιομηχανία είναι στρατηγική τομή της οικονομίας ε, που αξίζει τον κόπο μια πρωτοβουλία οικονομικής διπλωματίας. Ακούστηκαν ήδη, αλλά και οι μικρομεσαίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι και ελπιδοφόρες και, και κερδοφόρες και φέρνουν ανάπτυξη. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχει ανάπτυξη και στο εξωτερικό ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και εδώ απευθύνω έκκληση και προς την αριστερή πτέρυγα του Κοινοβουλίου να υποστηρίξετε το TTIP για να έχουμε καλύτερο πλαίσιο. Παγκόσμιες επαφές ε, για εξαγωγέ υπάρχουν ε, οργανισμοί προώθησης ε, εξαγωγών ε, στα κράτη-μέλη, διάφορα επιμελητήρια, αλλά μπορούμε και εμείς να κάνουμε περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, χρησιμοποιήσει περισσότερο τα παγκόσμια δίκτυα που διαθέτει και η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, οι διάφορες αντιπροσωπείες ακούστηκε, θα, πρέπει να, ή θα μπορούν να παίρνουν μαζί τους στις αποστολές και επιχειρηματίες. Λεφτά έχουμε στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και πολλά να διοργανώνουμε τέτοια πράγματα, να παίρνουμε μαζί μας επιχειρηματίες. Η Ευρώπη έχει δυνατότητα και θα πρέπει να τις αξιοποιεί ε, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, με τα κράτη-μέλη. Το παγκόσμιο εξαγωγικό εμπόριο θα πρέπει να διευκολυνθεί για τους μικρομεσαίους να ενισχυθεί και καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την πρωτοβουλία του κυρίου Ταγιάννη και να την εντείνει. Πολύ δε περισσότερο που οι εταιρείε μα στο εξωτερικό είναι και θετικός πρέσβης της ευρωπαϊκής ιδέας. Ευχαριστώ. Και πάλι για 1,5 λεπτό ο κύριος Σαλίνη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Πίτροπε. Η διάσταση της οικονομικής διπλωματίας ε, είναι ε, ουσιαστικά ολοκληρωμένο μέρος της φύσης της Υπήρου μας. Ε, οικονομικό πλαίσιο ήταν πάντα το πλαίσιο μέσω του οποίου η Ευρώπη αφηγήθηκε στον κόσμο ένα αναπτυξιακό μοντέλο ισχυρό, εύρωστο και βιώσιμο που βασίζεται σε μεγάλη δημιουργικότητα των επιχειρηματιών μας και των πολιτών μας αφενός και αφετέρου τη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός του ανθρώπου. Επομένως, δημιουργικότητα αλλά και ικανότητα οικοδόμησης ενός κοινωνικού μοντέλου. Για να κάνουμε όμως οικονομική διπλωματία θα πρέπει να γνωριζόμαστε καλά, να ξέρουμε σε τι είμαστε ισχυροί και να μπορούμε και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας για να τον προβάλλουμε. Εμεί είμαστε καλύτεροι στη μεταποίηση και δεν έχουμε πολλές πρώτες ύλες. Έτσι λοιπόν μια πρώτη στρατηγική στην οικοδόμηση πραγματικής οικονομικής διπλωματίας είναι να συνδέσουμε την παραγωγική μας ικανότητα με την δύναμη των χωρών που έχουν πρώτες ύλες και αυτά να συμβαδίζουν στη μεγάλη πρόκληση της Μεσογείου, μία πρόκληση εντός της οποίας η οικονομική μας διπλωματία μπορεί να διαδραματίσει εξαιρετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, μεγάλες σχέσεις και μεγάλες ικανότητες υποβολής προτάσεων, να προβαλόμαστε ε, και να υπερασπίζουμε τον εαυτό μας και να δημιουργήσουμε ε, κάποιους ε, ηγέτες, διπλωμάτες που να μπορούν να βοηθούν και τους επιχειρηματίες μας που μας έχουν εκπροσωπήσει παγκοσμίω. Ευχαριστώ η κυρία Σουίτσα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταγιάννη ε, για την πρωτοβουλία του να διατηρεί αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αυτή είναι μια νέα έννοια ε, πολύ γνωστή στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νέα για την Ένωση. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον κύριο Ταγιάννη. 24% του ΑΕΠ του παγκοσμίου είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά χρειαζόμαστε οικονομική διπλωματία. Θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο εξωτερικής πολιτικής. Και δεν νοείται εξωτερική πολιτική χωρίς οικονομική διπλωματία. Βεβαίως θα πρέπει όλα αυτά να τα συνδέουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίζεται και να ε, συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη, με τις εταιρείε μας, αλλά και με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αλλιώς δεν πρόκειται να διατηρήσουμε αυτό τον ηγετικό ρόλο που έχουμε στην παγκόσμια οικονομία. Φυσικά όλα αυτά για ποιον τα κάνουμε, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Χρειαζόμαστε όμως να διεθνοποιήσουμε την οικονομική διπλωματία και να εστιάσουμε πάρα πολύ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι ξέρουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα ποιοι είναι αυτοί. Αυτό είναι το ζήτημα. Στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν ήδη και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες και να εξάγουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής πριν το ΚΑΤΣΙΑ είναι ο κύριος Πόλτσακ. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αρχικά σκόπευα να ξεκινήσω διαφορετικά την ομιλία μου. Όλα τα άκουσα την ομιλία του Επιτρόπου, άλλαξα γνώμη και τώρα θέλω να σας θέσω μια ερώτηση. Ποιοι είναι οι στόχοι της οικονομικής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιστεύω ότι ο κύριος Επίτροπος το ανέφερε μερικώς. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω τα όσα είπε η κυρία Γκραπίνη, η οποία ρώτησε ποια συγκεκριμένα εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εκεί είναι η συγκεκριμένη στόχη της οικονομικής διπλωματίας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές και έτσι λοιπόν θα έπρεπε να διαδραματίσει και ισχυρότερο ρόλο σε διεθνές επίπεδο γενικότερα. Δεν έχουμε ισχυρή εκπροσώπηση ακόμη και υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα. Ο κύριος Σταγιάννη ανέφερε τρεις στόχους και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε περισσότερο τις επιχειρήσεις μας και τις εταιρείε μας γιατί ένα από τα κύρια επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχουμε μια καλή επιτυχή εταιρεία σε, στις διεθνείς αγορές. Αυτός θα πρέπει να είναι σε ένας από τους κύριους στόχους μας. Και αυτό είναι και ένα από του κύριου λόγου για να αναπτύξουμε την οικονομική διπλωματία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Έχω τέσσερι τώρα ομιλητέ και ομιλήτριε στο Catch the Eye. Θα σα δώσω το λόγο σε όλου. Ο κύριο Νότη Μαριά πρώτο. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με τις υπάρχουσες πολιτικέ δυνάμει, μια ευρωπαϊκή οικονομική διπλωματία θα εκπονείται και θα εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέτρα των γαλλογερμανικών θα παραμερίζει τους πολίτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ θα δεσμεύει τα κράτη με αποφάσεις που δεν ανταποκρίνονται στην ελεύθερη βούληση των πολιτών τους. η ιονή της οικονομικής διπλωματίας έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η επιτροπή είναι ακρο αρνητική για τους λαούς. οι καταστροφικές αποφάσεις λήψης μέτρων κατά της ρωσίας είχαν εξ αντιδιαστολής σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές επιχειρήσεις χωρίς μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή ένωση να έχει αποζημιώσει ικανοποιητικά και δίκαια τους πληγέντες ταυτόχρονα ενώ υπάρχουν διαρροές εγγράφων που αποδεικνύουν τις επαχθείς διατάξεις για το περιβάλλον που επεξεργάζεται η ttip η επιτροπή συνεχίζει το business as usual. αυτά τα γεγονότα καταδεικνύουν την τροπή που επιχειρούν να δώσουν στην οικονομική διπλωματία οι ευρωκράτες και που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία ενός οικονομικού νάτο μιας οικονομικής αναδίπλωσης στα πλαίσια της δύσης μιας υπόκληση στα υπερατλαντικά γεωγραφικά συμφέροντα που αγνοούν πλήρως τη λαϊκή ετιμιγορία και αποδεικνύουν επιδεικτικά ότι αγνοούν την, την πολυπολική συγκρότηση της παγκόσμιας οικονομίας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ιάκοφτσιτς. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Οικονομία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική και να αναπτυχθεί. Για να γίνει αυτό πρέπει να διεθνοποιηθεί ε, η οικονομία της, διότι το μερίδιο της ευρωπαϊκής οικονομίας συρρυκνούται όσο αναπτύσσεται και επεκτείνεται η παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία η οικονομική διπλωματία. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργειες με τις διπλωματίες των κρατών μελών σε πολλά κράτη-μέλη. Ε, και συνεργασία με χώρες της Νοτιοαμερικής και της Αφρικής. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή έτσι θα πρέπει να ειδωθεί και να συνδεθεί και με ένα άλλο θέμα, το οποίο επανέρχεται ξανά και ξανά και αυτό είναι το θέμα της μετανάστευσης που μας απασχολεί πάρα πολύ το μεταναστευτικό. Μπορούμε να το δούμε και με άλλο τρόπο στο σημερινό κόσμο η βιομηχανία, η ενέργεια είναι σημαντικά στοιχεία και για την οικονομική διπλωματία και ο τουρισμός. Θα πρέπει να οργανωθούμε όμως καλύτερα. Η κυρία Κονέτσινα έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Η οικονομική διπλωματία έχει συμφερόν να προωθήσει τους ευρωπαϊκούς οικονομικούς στόχους στο εξωτερικό. Η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά ισχυρίζονται ότι έχουν κατά νου τις μικρές και μισές επιχειρήσεις και όχι τις μεγάλες πολυεθνικές. Επίσης, ε, αναφέρεται και το θέμα της TTIP. Όμως ποια είναι η αλήθεια, μόνο το 30% των μικρών επιχειρήσεων εξάγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα πολύ κακό αποτέλεσμα της υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας και τις επιχειρήσεις μας με μεγαλύτερο σθένος. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις μικρές εταιρείες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις αλλοδαπές αγορές, όχι μόνο τις πολυεθνικές. Και πρέπει να πω κάτι στο συνάδελφο από το ΕΛΚ. Δεν χρειαζόμαστε τη ΣΥΤΑ και την τίτιπ, Θα πρέπει να έχουμε τάξη εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εδώ, αν δεν μπορούμε να οργανώσουμε τα πράγματα, δεν μπορούμε να το κάνουμε κι αλλού. Κύριε Ρούσα Τόμασιτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι αυτό που θέλουμε είναι να αναπτύξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομία, να προσελκύσουμε επενδύσεις. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή. Πολλά κράτη-μέλη έχουν το δικό τους μοντέλο οικονομικής διπλωματίας Και γιατί να μην ε, προωθούν και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στο εξωτερικό. Χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών ε, και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε ε, αυτή την προσπάθεια. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο θεσμικό αυτό και θεσμοθετημένο. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν πάντα τα ίδια συμφέροντα, ούτε τις ίδιες φιλοδοξίες. Η οικονομική διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βασικά ευνοεί τα πιο ισχυρά κράτη-μέλη βάρος των υπολείπων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατάινεν έχει τώρα το λόγο για να απαντήσει. Είναι και το ομιλητής για απόψε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τόσο καλή συζήτηση. Χαίρομαι πάρα πολύ Βλέπω τον κύριο Ταγιάννη ε, παρόντα, που ήταν και ο εμπνευστή ε, της οικονομικής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς λανσάρατε αυτή την ιδέα και αυτή την έννοια όταν ε, ήσασταν αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς φιλοδοξούμε να τη συνεχίσουμε και να τη μεταξελιξούμε για να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές οι διπλωματικές μας δραστηριότητες. Ετέθη μια καλή ερώτηση. Ποιοι είναι οι στόχοι της οικονομικής διπλωματίας. Προσπάθησα να εξηγήσω προηγουμένως τι κάνουμε. Και διευκρινίζουμε τους στόχους μας. Δηλαδή, δύο οικονομικούς διαλόγους υψηλού επίπεδου είχαμε με τρίτες χώρες. Πρώτον, με την Κίνα που συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς. Ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντώ το μάκαι αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ε, ε, με άλλους επιτρόπους βεβαίως και από κινέζικης πλευράς είναι και άλλοι αξιωματούχοι και υπουργοί. Στις συναντήσεις αυτές έχουμε και συζητήσεις καμιά φορά με τον ιδιωτικό τομέα Προσκαλούμε ιδιωτικέ εταιρείε να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο για να ακούμε και τις δικές τους απόψεις και τι περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τι περιμένουν από την την πλευρά την κινέζικη και ποιες είναι οι προτεραιότητες και τι μας ζητούν να κάνουμε εμείς για να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Την περασμένη φορά, το Σεπτέμβριο μάλιστα στο Πεκίνο, ο Επίτροπος Ότιγκερ συμμετείχε και η Επίτροπος Μπούλτς στις συζητήσεις αυτές και στο διάλογο και συζήτησαν θέματα συνεργασίας ε, για την πέμπτη γενεά, την τηλεφωνία πέμπτης γενεάς, το 5G. Και η Επίτροπος Μπούλς ε, μιλούσε για διασύνδεση διαφόρων πλατφορμών και ενδεχόμενες κινέζικες επενδύσεις στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα λοιπόν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την τεχνική μας βοήθεια ε, για τη χρηματοδότηση, ένα ταμείο ε, της, ε, του δρόμου του μεταξιού, το οποίο ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ευρώπη. Τέτοιου τύπου λοιπόν είναι ο διάλογος υψηλού επίπεδου που έχουμε με την Κίνα. Και πριν από λίγους μήνες, δύο μήνες, είχαμε αντίστοιχο διάλογο στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη με την Τουρκία. Με ε, αντιπροσωπείες επιχειρηματιών από την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση που συναντήθηκαν και μας έδωσαν και εκείνοι τις ιδέες τους για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κατέρωθεν ε, το εμπόριο και το επιχειρηματικό περιβάλλον και κλίμα. Και πάλι είχαμε τέτοιου τύπου συζητήσεις για την κανονιστική συνεργασία, για μακροοικονομικά ζητήματα. Ο Επίτροπος Μοσκοβισή επίσης παρευρέθη μιλήσαμε για συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη ε, με την Τουρκία. Μερικά μόνο παραδείγματα σας δίνω για τις τρέχουσες δραστηριότητές μας. Και αυτό δείχνει ξεκάθαρα ποιοι είναι οι στόχοι. Το είπα και προηγουμένως και ακούσαμε και από τη συζήτηση ότι ένας από τους τομείς προτεραιοτήτων είναι εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Πρέπει επίσης να αναφέρω την αναπτυξιακή πολιτική εδώ. Αναπτυξιακή βοήθεια και επενδύσεις. Εμπόριο και επενδυτική συνεργασία. Γιατί πολλές από τις χώρες της Τρίτης που βοηθούμε να αναπτυχθούν και να μεταρρυθμιστούν και είναι ε, αποδέκτες ε, αναπτυξιακής βοήθειας θέλουν να γίνουν εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι δικαιούχοι αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, εκεί υπάρχει χώρος ανάπτυξης και παίζει μεγάλο ρόλο οικονομική διπλωματία. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα είδος ταμείου, αντίστοιχο με αυτό που έχουμε με το ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που θα υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε τρίτες χώρες. Αυτή είναι μία από τις ιδέες μόνο. Τέλος. Να, να πω δύο λόγια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανέφερα ήδη τις εμπορικές συμφωνίες, αλλά πρέπει να προσθέσω και κάποια άλλα θέματα. Το ρόλο των ε, δικτύων των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών εμπορικών κλάδων σε τρίτες χώρες. Έχω γνωρίσει εξαιρετικά εμπορικά επιμελητήρια στην Κίνα, επί παραδείγματι. Είναι τα μάτια μας και τα αυτιά μας και παρακολουθούν τα τεκτενόμενα ε, καθημερινά στο εμπόριο στην Κίνα και στη Σιγκαπούρη επίσης όταν επισκέφθηκα και στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και στην Τουρκία. Και στο Ιράν επίσης που ακούστηκε προηγουμένως. Ε, αν όμως το Κοινοβούλιο έχει καλές ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ακόμα τη βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις ακούσουμε παρακαλώ. Μπορούμε να κάνουμε και εμπορικέ επισκέψει για υποστήριξη του εμπορίου και πρόθεση. Εκτό από την πρόθεση των εξαγωγών, μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο ας καινοτομήσουμε λίγο, ας ε, το πάρουμε αλλιώς, ε, να σκεφτούμε διαφορετικά. Um, Έχετε εμπειρία ε, στις συμβουλευτές και σε θέματα εμπορίου και σε θέματα προώθησης εμπορίου και η συμβουλή σας είναι πολύτιμη. Εγώ έχω ανοιχτό πνεύμα, να δεχτώ ότι μου πείτε, για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες να αναπτυχθούν και ε, τόσο το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Äh, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ